Um, um, Κυρίε και κύριοι, καλώς ήρθατε στη δεύτερη κοινή συνεδρία των Επιτροπών Εσωτερικής Αγοράς και Βιομηχανίας ε, στην οποία προεδρεύω μαζί με τον πρόεδρο Μπούζακ. Πρόκειται για την έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας προς μια νέα πράξη ενιαίας αγοράς. Το μόνο θέμα στην και διάταξη εγκρίνεται. Ωραία, οπότε να κάνω κάποιες ανακοινώσεις. Η συνεδρίαση μεταδίδεται στο διαδίκτυο. Υπάρχει διερμηνία σε όλες ε, τις γλώσσες πλην ε, μαλτέζικη σλοβακική και βουλγαρικής. Ορίστε. Και καλωσορίζω τα μέλη της Επιτροπής. Από την προηγούμενη συνεδρίασή μας είχαμε 1287 τροπολογίες που κατατέθηκαν χωρίς να μετράμε τις τροπολογίες ε, από τις νομοδοτήσεις των άλλων επιτροπών. Αυτό βεβαίως καταδεικνύει το τεράστιο ενδιαφέρον που υπάρχει από ανθρώπους από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο και παραπέρα. Ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ και συγχαίρουμε τους συνεισηγητές ε, Κάλας και Γκέπχαρτ. Είδα λοιπόν κάποια πρώτα σχέδια συμβιβαστικών τροπολογιών και ξέρω πως κάνετε πολύ σκληρή δουλειά για να προσπαθήσετε να βρείτε μια συμβιβαστική συμφωνία. Θα εγκριθεί η ε, Επιτροπή από κοινέ ε, συνεδριάσεις ε, που θα είναι πάντα υπό κοινή προεδρία των δύο προέδρων. Δύο ώρες προβλέπονται για αυτήν την συζήτηση. Εγώ θα προεδρεύσω στο πρώτο μέρος και μετά ο κύριος Μπουζεκ το δεύτερο θα ήθελα να σας ε, παρακαλέσω ε, αν, θέλετε το λόγο να το δηλώσετε σύντομα γιατί η γραμματεία θα προσπαθήσει να συγκεντρώσει τους ομιλητές. Οπότε μπορείτε να σηκώσετε το καρτελάκι σας μέχρι κάποιος να σας κάνει νόημα από τη γραμματεία. Και μετά, όταν θα φωνάξουμε το όνομά σας θα προσπαθήσουμε να τα μοιράσουμε μεταξύ των δύο επιτροπών και των πολιτικών ομάδων οπότε οι άλλες επιτροπές είναι απασχόλησης πολιτισμού και λίμπε θα δώσω λόγο στον κύριο Μπούζεκ να κάνει μια εισαγωγή και μετά θα ξεκινήσουμε την πρώτη ανταλλαγή. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε που είσαστε εδώ μαζί μας. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα πέραν του γεγονότος ότι ε, για τους εισηγητές και σκιώδεις δεν χρειάζεται να σηκώσουν τα χέρια τους γιατί θα πάρουν ε, αυτοδίκαια τον ε, λόγο. Εδώ νομίζω λοιπόν ότι ε, δημιουργούμε ένα πολύ καλό προηγούμενο αγαστή συνεργασίας μεταξύ επιτροπών και ε, δουλεύουμε από κοινού για την ε, ψηφιακή αγορά και την ενιαία ψηφιακή αγορά και νομίζω ότι δημιουργούμε ένα, μια καλή ομάδα, ένα κλάστερ κοινοβουλευτικών επιτροπών που θα μας δώσουν τη δυνατότητα να δούμε το θέμα αυτό από πολλές ε, πλευρές. Ε, ε, στην Κομισιόν έχει δημιουργηθεί ένα τέτοιο κλάστερ, μια τέτοια ομάδα ανάμεσα στον Πρόεδρο και τους αρμοδίους αντιπροέδρους και κάτι αντίστοιχο κάναμε και εμείς. Τώρα κυρία Πρόεδρε έχετε το λόγο. Να πω ίσως ότι Συναντηθήκαμε επίσης με τον Πρόεδρο και μέλη της Επιτροπής ε, ε, Πολιτισμού που είπαν ότι ενδεχομένως καλό θα ήταν ε, να σκεφτούμε τη διοργάνωση μιας ακρόασης για το geo-blocking, κοινής ακρόασης. Ο κύριος Κάλλας και η κυρία Γκέμπχαρτ. Ποιος, η κυρία Κάλλας και η κυρία Γκέμπχαρτ. Ποιος θα ξεκινήσει <laughs> πρώτος, η κυρία Κάλλας. Ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή σας. Δεν θα επαναλάβω το πόσες πολλές τροπολογίες έχουμε λάβει. Θα ήθελα βέβαια να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους που έδειξαν ενδιαφέρον για αυτό το ιδιαίτερα σημαντικό θέμα. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό το τι θα πει το Κοινοβούλιο στην έκθεση αυτή και τον τρόπο με τον οποίο ε, θα ε, προβλέψει ή θα αναφέρει την υλοποίηση της ψηφιακής στρατηγικής και της ε, ψηφιακής ενίας αγοράς θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τα χρονικά όρια έτσι ώστε να μπορέσουμε να επηρεάσουμε την διαδικασία στην Κομισιόν. Βεβαίως προσπαθούμε να ενσωματώσουμε όσο γίνεται περισσότερες τροπολογίες και όσο γίνεται περισσότερες προτεραιότητες. Ωστόσο ταυτόχρονα προσπαθούμε να κρατήσουμε την εστίαση ε, που πρέπει να έχει η έκθεση αυτή και να μην το στολίσουμε με υπερβολικά πολλά και να το κάνουμε τελικά χριστουγεννιάτικο δέντρο. Υπάρχουν πολλά που μπορούν να αναφερθούν ε, στο θέμα αυτό. Ε, πρόκειται για ε, ένα μεγάλο μέρος κεντρικό της ζωής μας το οποίο αναφέρεται στον ψηφιακό κόσμο <clears throat> και επομένως εμείς δίνουμε την δέουσα σημασία. Καταρχήν προσπαθούμε να δεχτούμε, να κάνουμε τέτοιες συμβιβαστικές τροπολογίες ώστε να παραμείνει απαράλλαχτη, ανέγγιχτη η δομή ε, της έκθεσης αλλά να δώσουμε όλα τα επιπλέον στοιχεία τα οποία χρειάζονται. Ε, επίσης ε, επενδύσεις, μάλλον όχι, το, το θέμα της ασφάλειας του κυβερνοχώρου είναι κάτι που έχουμε συζητήσει επανειλημμένα. <clears throat> Αλλά πρώτα θα ήθελα να πω δύο λόγια όσον αφορά τις τηλεπικοινωνίες. Είναι πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο ε, θα το, οποίο θα κινητροδοτεί τις ε, ιδιωτικές επενδύσεις. Ε, θα πρέπει να κρατήσουμε δηλαδή τον ανταγωνισμό ως κυρίαρχο στοιχείο των επενδύσεων λιγότεροι ε, operators, ε, ε, αν σε μια χώρα έχουμε λιγότερους operators, αυτό θα έχει ας πούμε κακή επίπτωση στους χρήστες. Επίσης, η ιδέα της ενδυνάμωσης του ρόλου του Μπέρεκ δεν είναι μια δημοφιλής ιδέα. Ωστόσο, το σημαντικό είναι να μην καταστή ο, ε, η παρούσα ρυθμιστική αρχή, αλλά να έχουμε μια συνολική εικόνα της ευρωπαϊκής αγοράς, γιατί μιλάμε για ουδετερότητα, η οποία θα πρέπει να αφορά το σύνολο της ευρωπαϊκής αγοράς. Ε, άρα κάποια επιπτεύουσα αρχή θα πρέπει να ε, υπάρχει που να ελέγχει ότι κάποιος δεν προσπαθεί να καρποθεί, ας πούμε, κάποια ωφέλη προς ζημία κάποιου άλλου. Αυτό το θέμα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό για την ε, Ήτρε και επομένως ε, χαιρόμαστε που υπάρχει γενικότερη στήριξη της πρότασης της Κομισιόν για ψηφιοποίηση της βιομηχανίας. Η καταγραφή των ε, η αρχή της, της καταγραφής ε, των δεδομένων ε, από τις δημόσιες υπηρεσίες. Αυτό είναι χαίρομαι γιατί αυτό ε, έχει βρει σύμφωνους πολλούς από τους συναδέλφους. Το e-government είναι πολύ σημαντικό οι τροπολογίες οι οποίες αναφέρονται σε ε, καινοτόμα οικοσυστήματα και κλάστερς ε, και την καινοτομία γενικότερα είναι πολύ σημαντικά. Οι ε, νεοφυείς επιχειρήσεις και μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι συχνά αυτές από τις οποίες ξεκινάει η καινοτομία. Για τα big data Ξέρουμε ότι δεν θα επενδύσουν σε αυτά οι μικρομεσαίες και οι νεοφυείς εάν δεν καταλάβουν ότι ε, και οι εθνικές αρχές και η Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύει ε, σε αυτά. Επίσης, ε, πολλές είναι οι τροπολογίες οι οποίες αναφέρονται στις πλατφόρμες και υπογραμμίζουν τις ε, διαφορές ε, ε, που υπάρχουν, την ποικιλία που υπάρχει στις πλατφόρμες. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε μία γενική και ίδια προσέγγιση για όλους. Η, ρύθμιση, η νομοθετική των πλατφορμών είναι σημαντική για τους πολίτες και για τους χρήστες. Πιστεύω επίσης ότι οι τροπολογίες οι οποίες εστιάζουν τις ε, υπηρεσίες που παρέχουν οι πάροχοι των ε, πλατφορμών είναι ε, θετικές. Από τις πλατφόρμες πηγαίνουμε στην sharing economy. Πολλές είναι οι τροπολογίες οι οποίες υπογραμμίζουν την ευκαιρία που έχει δώσει η sharing economy Ε, και την ανάγκη να ε, ε, δώσουμε μια νέα διάσταση σε αυτήν την sharing economy η οποία θα δώσει μεγαλύτερη δύναμη στους πολίτες και τους καταναλωτές. Αυτό που μας τρομάζει ας πούμε είναι ότι οι καταναλωτές οι καταναλωτές εμπιστεύονται όλο και περισσότερο τους άλλους καταναλωτές ε, και επομένως πολύ συχνά ε, ε, τις επιλογές τους τις κάνουν σύμφωνα με, τις, με τα σχόλια ή τις γνώμες άλλων χρηστών. Αυτό θα πρέπει να το δούμε. Μπορούμε να βρούμε βέβαια ένα τρόπο να το αναφέρουμε και να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να ρυθμίσουμε τις επιλογές ε, που μπορούν να κάνουν ε, οι ε, καταναλωτές. Αυτά ήθελα να πω και βεβαίως με πολύ θετικό βλέμμα κοιτάμε προς όλη αυτή τη συνεργασία που έγινε και προσδοκούμε και σε μελλοντική συνεργασία. Ευλίν Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω όλους τους ε, συναδέλφους που υπέβαλαν ε, τροπολογίες ε, που καλύπτουν ένα πραγματικό πραγματικά μεγάλο κομμάτι του κειμένου και είναι πάρα πολύ σημαντικό και ήταν εξ αρχής σαφές πως δεν μπορούσαμε να αναφερθούμε σε όλα τα θέματα γιατί δεν υπήρχε και αρκετός χώρος. Γι' αυτό θα είναι απολύτως ε, απαραίτητο, κυρία Κάλλας, και εδώ πέρα λίγο διαφωνούμε, να επιμηκυνθεί το κείμενο, γιατί ακριβώς έπρεπε να συμπεριλάβουμε αυτές τις ε, πτυχές, γιατί έπρεπε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχουμε μια ευρύτερη οπτική των πραγμάτων και να δούμε πώς θα μπορέσουμε να αναφέρουμε πράγματα τα οποία παραδείγματος χάρη δεν ανέφερε η Κομισιόν. Κάτι το οποίο οφείλουμε στους πολίτες να κάνουμε σοβαρή δουλειά. Γι' αυτό δεν θα ήθελα να περιοριστώ στον αριθμό εδαφίων κτλ και πολλές ε, τροπολογίες που καταθέσαμε νομίζω και κατατέθηκαν καταδεικνύουν ότι αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό το οποίο είναι γενικά θετικό είναι πως ε, δείχνουμε πως χρειάζεται μία θετική προσέγγιση του ψηφιακού κόσμου. Πρέπει δηλαδή να φροντίσουμε να έχουμε μια νέα προσέγγιση στην καινοτομία, τη δημιουργικότητα, τις ε, startups, να φροντίσουμε να εκμεταλλευτούμε όλες αυτές τις ευκαιρίες που μας δίνει ο ψηφιακός κόσμος. Υπάρχουν κάποια πράγματα στα οποία συμφωνούμε στο Κοινοβούλιο μεταξύ των οποίων η ουδετερότητα στο διαδίκτυο που μπορούμε να πούμε ξεκάθαρα πως έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα. Επίσης είναι ξεκάθαρο πως πρέπει να προχωρήσουμε σε ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων. Και από την άλλη δεν θέλω να κρύψω πως υπάρχουν κάποιοι τομείς που ακόμα τα συζητάμε. παραδείγματος χάρη, το θέμα, το, το θέμα των ε, τηλεπικοινωνιών όπου υπάρχουν ε, αρκετές διαφορετικές απόψεις ε, το θέμα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με την αρχή ότι κάτι γίνεται άπαξ και διαπαντός και να δούμε άρα το τι μπορούμε να δεχτούμε και το τι όχι νομίζω πως πρέπει να τα συζητήσουμε αυτό να τα συζητήσουμε αυτό το ζήτημα. επίσης το θέμα του δικαίου των ε, συμβάσεων. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, ε, στις οποίες θα πρέπει να εμβαθύνουμε και βέβαια αναμένω να δω τι θα μας πει και η Κομισιόν και βεβαίως ε, να δούμε το τι θα κάνουμε με την οδηγία των υπηρεσιών. Υπάρχουν αυτοί που λένε ότι πρέπει να τις ξανανοίξουμε, δεν θεωρώ πως είναι αυτή η σωστή προσέγγιση θα πρέπει κάποτε να δούμε την εφαρμογή του υφιστάμενου δικαίου στα κράτη-μέλη πριν κάνουμε κάτι το καινούριο. Δεν έχει νόημα να λέμε θα κάνουμε κάτι καινούριο αν δεν έχει εφαρμοστεί το παλιό. Και πρέπει στο πλαίσιο αυτό να σκεφτούμε τι θα κάνουμε στους ε, τομείς αυτούς ε, όσον αφορά την ίδια κριτική μεταχείριση στις υπηρεσίες ή να το δούμε και στο πλαίσιο του ανταγωνισμού. Θεωρώ πως ε, θα πρέπει να τα δούμε όλα αυτά. Μετά υπάρχει το θέμα των διαφόρων ε, πλατφορμών. Εδώ πέρα συμφωνούμε με την κυρία Κάλλας. Υπάρχουν διάφορες πλατφόρμες και μορφές τέτοιων πλατφορμών δεν μπορούμε να δώσουμε έναν ενιαίο ορισμό γιατί αφορούν και υπηρεσίες ε, που προσφέρονται ε, είτε μιλάμε για μηχανές αναζήτησης ή υπηρεσίες όπως ε, το Uber ή Clickworking για να αναφέρω δηλαδή τρεις τελείως διαφορετικές πλατφόρμες γι' αυτό πρέπει να σκεφτούμε τι θα κάνουμε σε αυτούς τους ε, τομείς και εδώ πέρα νομίζω πως υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να επεξεργαστούμε και το οποίο δεν υπάρχει σε αυτά τα οποία μας πρότεινε η Κομισιόν η αξιολόγηση αντικτύπου στην κοινωνική ζωή, στην εργασιακή ζωή των πολιτών, στην κοινωνία την ίδια. Δεν το βλέπουμε αυτό στην πρόταση της Κομισιόν. Βεβαίω δεν μπορούμε να κοιτάμε μόνο τις, κοινων... τις οικονομικές πτυχές ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να αγνοούμε τους πολίτες χωρίς τους οποίους δεν θα υπάρξει κάποια επιτυχία τους πολίτες και τα κοινωνικά τους δικαιώματα. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε μια μεγαλύτερη έμφαση σε αυτό. Γιατί εγώ πάντα έλεγα και το είχα πει και στην οδηγία υπηρεσιών ότι η οικονομική πολιτική αφενός και η κοινωνική πολιτική η αφετέρου δεν είναι πράγματα αντιφαντικά. Μόνο εάν τα συντεριάξουμε μπορούμε να προωθήσουμε την κοινωνία οτιδήποτε άλλο πραγματικά θα πρόδιδε τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναμένω τι έχουν να πούν οι συνάδελφοι. So the next speakers will each have uh, minutes each, going through the... Τρία λεπτά έκαστος ε, για τις πολιτικές ομάδες, ε, ε, οι σκιώδες δηλαδή, από τις επιτροπές Ένα Φεκούχαν. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις ε, συνεισηγήτρες ε, Κάλασε και Κέφχαρτ, λέει η κυρία Βερκούνεν, ε, για τη δουλειά που έχουν κάνει. Έχουν γίνει πάρα πολλά. Είμαστε ιδιαίτερα απασχολημένοι όλοι με τις τροπολογίες και τις συμβαστικές, οποίες θα καταλήξουμε τις επόμενες εβδομάδες. Θα ήθελα να τονίσω κάποια πράγματα για τα οποία επιμένει η πολιτική μας ομάδα. Από πλευρά τη ΣΥΤΡΕ καταρχάς καταθέσαμε τροπολογίες με τρόπο ώστε να ενισχυθεί η βιομηχανική ούτως υπήν βάση της έκθεσης, όπως είπε και η κυρία Καλές, επιταχύνοντας την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας, δημιουργούμε τις απαιτούμενες συνθήκες για την τόνωση της ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας είναι ένα από τα πράγματα στα οποία πρέπει να επικεντρωθούμε πώς ε, να τονώσουμε τη δημιουργία θέσεων εργασίας μέσω της ψηφιοποίησης. Ε, πώς να τονώσουμε την ανάπτυξη χάρη στην ψηφιοποίηση. Είναι σημαντικό. Ε, για την παραδοσιακή βιομηχανία, την μεταποιητική, τις μεταφορές, ε, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις δημόσιες υπηρεσίες, την παιδεία και εκεί θα πρέπει να δούμε ποιος θα είναι ο αντίκτυπος ε, της ψηφιοποίησης. Αντίστροφα, πώς μπορεί την ψηφιοποίηση να την τονώσει η ίδια η βιομηχανία, δηλαδή νέα μοντέλα, νέες υπηρεσίες, παραγωγικά μοντέλα, νέες υπηρεσίες να δημιουργηθούν, όπως βλέπουμε και σε άλλες τροπολογίες και του ΕΛΚΑ, διότι μιλάμε και για τον κανονισμό. Έχουμε ήδη πει ότι επιγραμμικά είναι σημαντικό να υπάρχει εμπιστοσύνη. Θα πρέπει όμως να μην είναι υπερβολικές οι ρυθμίσεις. Χρειαζόμαστε μεταρρυθμίσεις, ούτως ώστε να είναι πραγματική ενιαία ψηφιακή αγορά και για να συμβεί αυτό, να περάσουμε στην ψηφιακή εποχή, θα πρέπει να προσέξουμε να μην να αυξήσουμε υπερβολικά τις νομοθετικές ρυθμίσεις και το διοικητικό άχθος για τις επιχειρήσεις. Το αντίθετο πρέπει να κάνουμε. Ε, με την ε, ε, εναρμόνιση που επιδιώκουμε θα πρέπει να αντικαταστήσουμε την πεπαλαιωμένη, την παροχημένη νομοθεσία και όχι να προσθέσουμε ρυθμίσεις υφιστάμενες. Είναι μεγάλη πρόκληση αυτή για τα κράτη-μέλη. Κάτι άλλο. ψηφιακά αγαθά και υπηρεσίες. Ο ψηφιακός κόσμος φαίνεται να απέχει ορισμένε φορές από τον παραδοσιακό. Όμως ε, τα ψηφιακά αγαθά και υπηρεσίες πρέπει να την χάνουν ε, αντίστοιχες μεταχείρισης όπως για τα παραδοσιακά και ο κανονισμός θα πρέπει να καλύπτει το περιεχόμενο είτε είναι ψηφιακό είτε όχι. Σε αυτό επιμένουμε. Θέλουμε να υπάγονται στον ίδιο κανονισμό είναι μία από τι βασικές προκλήσεις ε, για το μέλλον. Περιμένουμε με ανυπομονησία τα αποτελέσματα της συνεργασίας με τους, ε, τις συνεισηγήτριες και όλους τους όλους εισηγητές είναι πολύ καλή η βάση και θέλουμε να την εμπλουτίσουμε την περαιτέρω την έκθεση. Ευχαριστούμε, Φιλίπ Ζου. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο εισηγητές ε, για την ευφυή εργασία την οποία έχουν ε, κάνει μέχρι τώρα. Έχουμε συναντηθεί πολλές φορές για το ίδιο θέμα, γι' αυτό θα ήθελα να μου επιτρέψετε να επιστήσω την προσοχή όλων ότι το θέμα είναι πολύ τεχνικό και είναι δύσκολο ε, να το δουλέψουμε. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να σας ζητήσω ε, έγκαιρα να έχουμε τις τροπολογίες ε, λιγότερο από 24 ώρες για να συγκρίνουμε εκατοντάδες τροπολογίες με συμβιβαστικές τροπολογίες. Γίνεται μία φορά αλλά όχι και συνέχεια. Όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών και πάνω σε πολλά άλλα πράγματα πολλά θα είχαμε να πούμε. Αλλά να συγκρατήσουμε ότι θα πρέπει στην έκθεση έκθεση, από την έκθεση να προκύπτει σαφώ ότι η ψηφιακή αγορά, ο ψηφιακό κόσμος δεν είναι κίνδυνο, αυτό θα πρέπει να είναι ο γενικό τόνο ε, τη έκθεση. Δεύτερον, το πιο σημαντικό είναι να δώσουμε ε, την ε, απαραίτητη εμπιστοσύνη που πρέπει να έχει ο καταναλωτής στο ψηφιακό κόσμο. Επομένως, ο καταναλωτής θα πρέπει να προστατεύεται με τον ίδιο τρόπο όταν αγοράζει κάτι επιγραμμικά ή κάτι σε ένα μαγαζί. Επίσης χρειαζόμαστε προστατευτικό νομοθετικό ε, ε, ε, πλαίσιο για την πώληση περιεχομένου επιγραμμικά. Όσον αφορά τώρα ε, την ε, πώληση προϊόντων ε, στο μέσο ίντερνετ, νομίζω ότι σκόπιμο είναι να πούμε ότι περιμένουμε τα αποτελέσματα της Refit για την προστασία των καταναλωτών και βεβαίως θα πρέπει η Κομισιόν πριν νομοθετήσει να ακούσει προσεκτικά και τη γνώμη μας. Επιμένω σε αυτό. Προστασία του καταναλωτή επίσης επίσης περνάει και μέσα από το geo-blocking και ευχαριστώ όλους όσοι ε, αναφέρθηκαν σε αυτό ε, geo-blocking το οποίο βεβαίως θα βασίζεται σε μια ισοδίκαιη κατανομή ε, του, της επικράτειας γιατί αυτά που ακούμε και τέτοιες λύσεις που ακούγονται είναι απαράδεκτες. Επίσης νομίζω ότι θα πρέπει να ε, ε, παρακολουθήσουμε τη θέση της Κομισιόν όσον αφορά ε, την, το round που ξεκίνησε στις 26 Μαρτίου του 2015 για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Επίσης, θα πρέπει να βοηθήσουμε τους καταναλωτές να ελέγξουμε τους παρόχους αλλά, χωρίς, αλλά διασφαλίζοντας ταυτοχρόνως και την εδαφική ισορροπία. Ε, αυτά θα είχα και πολλά άλλα να πω, αλλά σας ευχαριστώ πάρα πολύ ε, και επιμένω ότι όπως είπα και προηγουμένως οι συμβαστικές τροπολογίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ευχαριστώ πολύ. Μία πέτρα κομπούλα μάτρη. Ευχαριστώ. Και εγώ χαίρομαι για το θέμα αυτό. Χθες είχαμε μια συζήτηση στην ομάδα. Στην αρχή είχα απογοητευτεί για το ότι υπήρχε αυτή η έλλειψη ψηφιοποίηση στη βιομηχανία, αλλά πλέον μπαίνει και αυτό σιγά σιγά στην έκθεση και άρα νομίζω πως είναι κάτι στο οποίο μπορεί να μας ε, βοηθήσει η τρία. αλλά δεν πρέπει να περιοριστούμε μόνο στην ε, εσωτερική ενιαία αγορά πρέπει να κάνει περισσότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να συμφωνήσουμε πως η ψηφιακή αλλαγή είναι κοινωνική αλλαγή γιατί να μην αναφέρουμε ότι θα επηρεάσει την κοινωνία. Να μην πούμε ότι πρέπει να προετοιμαστούμε, να συζητήσουμε το ζήτημα αυτό σε πανευρωπαϊκό φόρουμ ή οτιδήποτε άλλο χρειάζεται. Ε, εμένα δεν με πείθει το ότι πρέπει να δούμε μόνο ε, τα 2016 και τα υπόλοιπα τα αφήσουμε. Δεν χρειάζεται να έχουμε τις απαντήσεις ε, μέχρι το 2016, αλλά ας ε, δείξουμε τουλάχιστον ότι ζούμε στο σήμερα. Επίσης, κάτι άλλο. Εντάξει, δεν μιλάμε για κβαντομηχανική και τα λοιπά αλλά θα πρέπει πράγματι να δούμε το ψηφιακό χάσμα το οποίο για εμάς είναι απαράδεκτο πρέπει να υπάρχουν επενδύσεις ε, στις υποδομές ε, από τις εταιρείες που θα πρέπει να στηρίξουν τα ευρωπαϊκά ταμεία αλλά έχουμε και πολλές ιδέες για το πώς μπορεί να γίνει αυτό χωρίς δημόσια χρηματοδότηση έτσι ώστε οι ευρωπαϊκές εταιρείες να μπορέσουν να ενταχθούν σε μια ηλεκτρονική κοινωνία. Έτσι θα μπορέσουν να ανθίσουν και η Εύελιν επίσης ανέφερε κάποια πράγματα αλλά υπάρχει και η οδηγία περί υπηρεσιών που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όσον αφορά τώρα τις πλατφόρμες δεν ανάγκη να έχουμε ένα μέγεθος για όλους, αλλά θα πρέπει να αποτρέψουμε τα μονοπόλια. Αν έχουμε, κάτι, αν έχουμε λόγο στην εσωτερική αγορά, πρέπει να μην έχουμε μονοπόλια. Δεν είναι η οικονομία της αγοράς με έναν ή δύο, δηλαδή iOS και Android αυτή τη στιγμή είναι 92% της αγοράς. Αν σε μπλοκάρουν αυτοί, δεν έχεις ψηφιακές λύσεις. Και βεβαίως δεν πρέπει να δούμε το τι κάνουν η της ε, στην ομοθεσία για τις ε, λοιπές ε, υπηρεσίες. Τώρα, είπαμε ότι θα είναι και μια κοινωνική επανάσταση. Θα θέλαμε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να δει τι θα γίνει με την πέμπτη γενιά κίνητης τηλεφωνίας και με τα υπόλοιπα. και ελπίζω όπως είπα να μεταδοθεί για πρώτη φορά σε 5G ένας αγώνας ποδοσφαίρου στην Ευρώπη και όχι στην Ασία. Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Αναμένω λοιπόν την επόμενη συζήτηση την Πέμπτη και άλλοι βουλευτές τόνισαν τις ευκαιρίες που προσφέρει η ψηφιακή ενιαία αγορά για επιχειρήσεις και καταναλωτές και θα ήθελα να δω λοιπόν και εγώ μια, ένα θετικό τόνο σε αυτή την έκθεση. Τώρα η κυρία Γκέπχαρτ πράγματι πρέπει να δούμε την υφιστάμενη οδηγία για τις ε, υπηρεσίες ε, να εφαρμοστεί όπου χρειάζονται αλλαγέ πρέπει να είναι στοχευμένες ε, προσεκτικά και να φροντίσουμε η νομοθεσία να αντέξει στις μελλοντικές εξελίξεις θα πρέπει να ξαναδούμε Επίσης ε, και του χρόνου, όπως είπατε, την ε, αναδιατύπωση και κωδικοποίηση της νομοθεσίας. Και βέβαια αναγνωρίζουμε πως ε, τα ψηφιακά αγαθά διαφέρουν από τα απτά αγαθά. Αν λείπουν παραδείγματο χάρη 12 σελίδε από ένα κανονικό βιβλίο μου, χρειάζεται ένα καινούριο βιβλίο, ενώ δεν ισχύει το ίδιο για ένα ψηφιακό βιβλίο. Επίση υπάρχει το θέμα της ε, παράδοσης ε, των ε, της παράδοσης σε κομμάτια αλλά και βεβαίως των ταχυδρομικών υπηρεσιών οι οποίες διαφέρουν πολύ από χώρα σε χώρα υπάρχει βεβαίως και το πακέτο που συζητάμε με τον Επίτροπο Έτιγκερ αλλά και τα δικαιώματα των καταναλωτών όσον αφορά τώρα τις εκκλήσεις που υπάρχουν για μια εναρμονισμένη πολιτική του φάσματος πράγματι πρέπει να το δούμε αυτό με τα κράτη-μέλη αλλιώς δεν γίνεται τίποτα οπότε θα μας βοηθούσε το Συμβούλιο να συνεργαστεί μαζί μας δεν συμφωνώ τώρα να έχουμε ε, μια ενιαία ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή τηλεπικοινωνιών κυρίως γιατί δεν έχουμε ευρωπαϊκά μονοπόλια. Υπάρχει ο Μπέρικ λοιπόν, ο οποίος έχει λάβει κάποιες περισσότερες αρμοδιότητες, αλλά δεν βλέπω κάτι. Τώρα η τυποποίηση είναι ένα ζήτημα για πολλές ομάδες. Χαίρομαι πως όλοι ανησυχούμε για τον κίνδυνο δημιουργίας μονοπωλίων. Δεν υποστηρίζω εγώ την ανοιχτή πρόσβαση άνευ ορίων Όσον αφορά τώρα τις πλατφόρμες, ούτε εκεί πέρα υπάρχει μία λύση για όλους. Συμφωνώ εδώ πέρα και υπάρχει και μία μεγάλη διαφορά στην συμμετοχική οικονομία. Εγώ θεωρώ πως αυξάνεται αυτή η οικονομία γιατί αρέσει στους καταναλωτές, αισθάνονται ότι έχουν κάποια δύναμη και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί να μην ε, ρυθμίσουμε τον κλάδο υπερβολικά, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να είναι ίση η όρη μου Ξέρω πως τα ζητήματα εργατικής νομοθεσίας και φορολογίας είναι εθνικό ζήτημα. Τώρα για το GDPR και το ασφαλή λιμένα πρέπει να βρεθεί ένας συμβιβασμός και υποστηρίζω και τις τροπολογίες που λένε πως το σύστημα GSM πρέπει να είναι προσβάσιμο σε άτομα με αναπηρία. Λοιπόν, ο Hans όλα λείπει για το ECR, οπότε Dieter για Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Με τόσες πολλές τροπολογίες δεν θα γινόταν τόσο να τις σχολιάσω όλες μεμονωμένα. Θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις από τη δική μας προοπτική. Το φαινόμενο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Το ανέφερε κάποιος. Ε, και συμφωνώ, συμφωνώ με αυτήν την επιθυμία που υπάρχει να τους ευχαριστούμε όλους, όμως ε, με ε, πάνω από χίλιες τροπολογίες είναι πλέον απαράδεκτο αυτό. Δηλαδή, εάν κάποιες τροπολογίες απλώς επαναλαμβάνουν σε πολλές διαφορετικές παραγράφους την ίδια δήλωση και είναι επαναλαμβανόμενες, θα πρέπει να περιοριστούμε γιατί κανείς δεν θα το διαβάσει το χριστουγεννιάτικό μας δέντρο ε, στο κάτω-κάτω της γραφής. Δεύτερον, ε, χρονοδιάγραμμα. Ε, μία από τι βασικέ προτεραιότητε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η ψηφιακή ενιαία αγορά. Οπότε ε, θα έπρεπε βασική προτεραιότητα δική μα είναι να περάσουμε αυτό το μήνυμα ότι είμαστε σε θέση για αυτό το θέμα προτεραιότητα να έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Κυρίω δεν πρέπει να δώσουμε την εντύπωση με αυτή την έκθεση ότι θέλουμε να επιβραδύνουμε την διαδικασία ολοκλήρωσης ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Αυτό θα είναι βασική προτεραιότητα για μας. Ε, τρίτον, δεν θα μπορέσουμε να δεχτούμε τις τροπολογίες που ως στόχο έχουν να προστατεύσουν τους παραδοσιακούς παρόχους μέσω νομοθεσίας ή ε, εμποδίζοντας την συνεργατική οικονομία με, με επιπλέον διοικητικό άκθο ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο για την ε, κοινωνική προστασία νομίζω ότι δεν είναι αυτός ο τρόπος ε, ε, να βελτιώσουμε τη ζωή των πολιτών, δηλαδή ισχυριζόμενοι, αρνούμενοι την ψηφιακή επανάσταση ή λέγοντας ότι χρειαζόμαστε νέα, τεχνη, νέους τεχνητούς φραγμούς για τον ανταγωνισμό προωθώντας μόνο τις παραδοσιακές βιομηχανίες. Θέλουμε να δώσουμε όθηση στη νέα ψηφιακή επανάσταση και γι' αυτό οι δικές μας τεχνολογίες είναι μελλοντοστραφείς και υπέρ της καινοτομίας. Αυτά θα βρείτε στις δικές μας τροπολογίες, νέες ιδέες, περιορισμός της απώλειας χρόνου λόγω διοικητικών διαδικασιών, υποστήριξη του ιδιωτικού τομέα, ώστε να είναι ανταγωνιστικό σε παγκόσμια κλίμακα. Χρειαζόμαστε μια ψηφιακή ενιαία αγορά όπου κερδίζουν οι καλύτερες ιδέες. Από όπου και αν έρχονται από ε, μία startup επιχείρηση ή από ε, την κυβέρνηση. Αυτά θέλω, αυτές οι ιδέες, οι βασικές ιδέες μας θέλω να πηχούνται στις, τροπολογίες, ε, στις συμβαστικές τροπολογίες τις οποίες τελικά θα καταλήξουμε. Η Κορνέλια Έρνεστ. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Ναι, να προωθήσουμε τον ανταγωνισμό. Εδώ πέρα συμφωνούμε. Αλλά αυτό το οποίο πρέπει να συζητήσουμε είναι η ισορροπία μεταξύ ανταγωνισμού και διαφύλαξης των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αν προσανατολιζόμαστε μόνο στον ανταγωνισμό, όσο σημαντικός και αν είναι, τότε έχουμε κάνει μόνο τη μισή δουλειά. Γι' είναι σημαντικό να δούμε και ζητήματα των ευκαιριών αλλά και των κινδύνων. Δεν έχει νόημα να, γράφουμε και να λέμε πράγματα και να, τα οποία στόχο έχουν μόνο να φρενάρουν αλλά το θέμα των προσωπικών δεδομένων είναι τεράστιο. Είναι επιχείρηση ξεχωριστή στην ψηφιακή οικονομία και θα πρέπει ακριβώς να αποκατασταθεί αυτή η ισορροπία. Το άλλο. Πρέπει ήρεμα να δούμε τι πρέπει να ρυθμίσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τι όχι. Να το δούμε αυτό προσεκτικά όχι να βάλουμε υπερβολικούς κανόνες για να κάνουμε πράγματα τα οποία θα είναι τελικά αντιπαραγωγικά. Γι' αυτό θεωρώ σημαντικό να έχουμε μια πολιτική φιλική στην καινοτομία οπωσδήποτε, αλλά χρειάζεται και προστασία δεδομένων από τον σχεδιασμό και εξορισμό. Πρέπει δηλαδή να είναι κάτι το ενσωματωμένο στην τεχνολογία. Και οι ρυθμίσεις για τους χρήστες να είναι έτσι ώστε εξορισμού να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα. Μετά μιλήσατε για μονοπόλια που δεν θέμε κτλ. Δεν είναι αδιάφορο το να υπάρχει ένα μονοπόλιο. Χρειάζεται πράγματι ποικιλομορφία. Πρέπει να μιλήσουμε για το δωρεάν software θεωρώ πως είναι μια σημαντική στιγμή. Και το τελευταίο, ο αποκλεισμό ε, που αναφέρθηκε. Πρέπει να γίνει κάποια ακρόαση για να δούμε σοβαρά το τι θα κάνουμε μεταξύ των τριών επιτροπών ε, ΕΚΟ, ΙΤΡΕ και ΚΟΥΛΤ. ΚΟΥΛΤ, ναι. Υπάρχουν λοιπόν ε, κάποια πράγματα που είναι άσαφη Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να είμαστε ήρεμοι. Δεν είναι ότι θα τελειώσει ο χρόνος. Εντάξει, να κινηθούμε σωστά, αλλά να μην ε, κάνουμε τα πράγματα τσαπατσούλικα. Ευχαριστώ. Υποθέτω ότι για την ε, γεωφραγή θα έχει και η Γιούρη να μας πει κάτι. Ο Ντένις Δε δεν είναι εδώ. Εάν δεν έχετε ήδη υποδείξει την επιθυμία σας να μιλήσετε στον επόμενο γύρο, παρακαλώ να το κάνετε τώρα, γιατί φαντάζομαι θέλουν κάποιοι. Ευχαριστώ τους συμπροεδρεύοντες. Εγώ χαίρομαι που ζήτησα το λόγο, διότι από πλευράς των Πρασίνων υποτίθεται παρότι εγώ δεν είμαι σε, ανήκω σε πρασίνων, αντικαθιστώ την Γιούλια Ρέντα. Ποιο μπορεί να αντικαταστήσει τη Γιούλια Ρέντα, τέλος πάντων. Μου ζήτησε να σχολιάσω κάποια ζητήματα και θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο και περιεκτικός. Τώρα τι να ευχαριστώ τις ε, συνεισηγήτρες, ξέρετε ότι με ευγνώμων, ας περάσω στο ψαχνό. Το geo-blocking θα πρέπει να καλύπτεται με όσο δυνατόν λιγότερε εξαιρέσει ε, γίνεται και η διάκριση λόγω γεωγραφικής ε, τοποθεσίας αντιβαίνει στην ίδια την αρχή ε, της ψηφιακή ενέργεια αγοράς και οδηγεί σε κατάτμιση της αγοράς. Επίσης, ε, για τα δικαιώματα των καταναλωτών, είτε επιγραμμικά είτε όχι, θα πρέπει να προσαρμόσουμε τις νομοθετικές ρυθμίσεις ε, πλέον. Δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία διακριτική μεταχείριση και κανένας καταναλωτής δεν θα πρέπει να έχει χαμηλότερο επίπεδο προστασία σε σχέση με αυτό που έχει τώρα. Μόνο και μόνο επειδή είναι ε, ψηφιακά τα αγαθά και οι υπηρεσίες. Τρίτον, Ω συνήθω ανησυχούμε γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι ξεκάθαρη για τον ορισμό που δίνει για τις πλατφόρμες. Αυτό θα έχει επιζήμιο αποτέλεσμα στις προσπάθειες που κάνουμε να είμαστε καινοτόμοι. Δεν μπορούμε να παραμείνουμε στην επιφάνεια, θα πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι και να κάνουμε ειδικότερα σχόλια. Τα ηλεκτρονικά βιβλία θα πρέπει να διαβάζονται όπως τα έντυπα. Να καλύπτονται λοιπόν από το δίκαιο πολίσεων για τα αγαθά και όχι για τις υπηρεσίες. Επίσης, ε, καμία διακριτική μεταχείριση σε σχέση με τις εξαιρέσεις ΦΠΑ. Εάν ε, το περιεχόμενο εξαιρείται, τότε η εξαίρεση θα πρέπει σε όλες τις μορφές ε, άειλες και υλικές να εφαρμόζεται, να μην υπάρχει καμία διακριτική μεταχείριση. Η πρόσβαση για τα αμαία, κυρίως όταν μιλάμε για την διασυνδεσιμότητα και όταν λέω σε, αυτό, σε αυτά τα συμφραζόμενα διασυνδεσιμότητα θα εννοώ συμβατότητα έτσι, για τα άτομα με ειδικέ ανάγκες. Ξέρουμε όλοι τι προβλήματα υπάρχουν. Κλείνοντας, να κλείσω με κάποιες ε, ευχές και επιθυμίες. Κάποιοι συνάδελφοι σχολίασαν ε, το φαινόμενο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Δεν μπορούμε να βάλουμε δωράκια για όλους κάτω από το δέντρο για να χαρούν όλοι. Και εγώ θέλω να προτείνω το εξή. Είναι πράσινο εξορισμού το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Οπότε να υιοθετήσετε τι προτάσει των πρασίνων και αφήστε τα υπόλοιπα υπό, απ' έξω. Μα είστε ε, αυτοδικαίως σκιώδης σε βάση του καταλόγου μου και η Γιούλια ε, ε, είναι επίσης σκιώδης. Θέλετε να πείτε και δικά σας ή θα μιλήσετε μόνο για τη Γιούλια. Το Τα περί χριστουγεννιάτικου δέντρου ήταν δικά μου σχόλια. Πολύ ωραία. David Μπορέλη. For the e And then I have Marco Και μετά ο Μάρκο Ζούλο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τις εισηγήτριες και τις γραμματείες τις αντίστοιχες οι οποίες ε, κάνουν επίπονη εργασία λόγω της περιπλοκότητας ε, του θέματος και λόγω της ε, κοινή εργασίας θα ήθελα να εστιάσω την προσοχή μου στην προσέγγιση που έχουμε. Η αρχική προσέγγιση των εισηγητριών αναμφισβήτητα ήταν η προστασία των πολιτών και των καταναλωτών και από αυτού μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι. Ε, σε γενικές γραμμές. Όσον αφορά τις αρχές, ε, φαίνεται ότι έχει προωθηθεί κι άλλο. Τα προβλήματα, κατά την άποψή μας, ε, προκύπτουν όταν από τις αρχές περνάμε στα συγκεκριμένα σημεία. Γιατί σε αυτήν την έκθεση πιστεύουμε ότι υπάρχουν στοιχεία αναντίστοιχα από τη μία πλευρά έχουμε το θέμα των ε, προτύπων ε, συμβάσεων. Έχουμε προβλήματα όσον αφορά τις διατυπώσεις οι οποίες μπορεί να είναι αντιφατικές. Αναφέρομαι ας πούμε στο geo-blocking όταν ε, μιλάμε στα πλαίσια του geo-blocking μια, για μια θετική διακριτική μεταχείριση. Αυτό είναι contradiction in terminis. Δεν είναι δυνατόν πάση θυσία να θέλουμε κοινή συνένεση ε, ή δεν μπορούμε να ευχαριστήσουμε λίγο όλους έτσι ώστε ε, ε, τελικά να τύχει μεγάλη έγκρισης ενδεχομένως η δεν μπορουμε να ευχαριστησουμε λιγο ολους ετσι ωστε τελικα να τυχει μεγαλη έγκριση ενδεχομενως Η εκκλησια η προσέγγιση κινδυνεύει να οδηγήσει σε ένα ασαφές αντιφατικό ε, κείμενο το οποίο θα μπορούσε να δημιουργήσει μεγαλύτερη σύγχυση. Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω τις ε, εισηγήτριες ε, να ακολουθήσουν αυτή την αρχική ιδέα για ένα κείμενο φιλόδοξο για ένα κείμενο καινοτόμο. Ε, οι ε, πολίτες θέλουν μια ε, ψηφιακή οικονομία η οποία θα βασίζεται πραγματικά στους τρεις σημαντικούς πυλώνες, συμμετοχή, οικονομία και εμπιστοσύνη. Ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο στον τελευταίο ομιλητή του πρώτου γύρου, να σας πω να δούμε λίγο τον κατάλογο. Griffin, Nielsen, Blanco Lopez, Thun, Uh, λοιπόν, εάν δεν ακούσατε το όνομά σας σε αυτό το... Ε, θα πρέπει να ζητήσετε το λόγο αν δεν ακούσατε λοιπόν το όνομά σας. Ε. Ε, άκουσα ε, κάποιους ε, να λένε μήπως να αργήσουμε λίγο, καθυστερήσουμε την ψηφοφορία για να κάνουμε ένα hearing, να οργανώσουμε ακρόαση. Όχι, όχι, δεν είναι δυνατόν. Αυτή είναι η δυνατότητα που έχει το Κοινοβούλιο να προωθήσει τις θέσεις του μέσα από γνωμοδότης τεσσάρων επιτροπών. Επομένως όλα αυτά θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί. Έχουμε συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια και δεν θα ήταν καλό να μην τα λάβουμε υπόψη μας. Από εκεί και πέρα, στην πρόθεση της νομοθετικής διαδικασίας θα μπορούσαμε να καλέσουμε εμπειρογνώμονες κτλ. Αλλά αυτό μπορεί να γίνει παρεπιπτόντος. Τελευταίος ομιλητής ε, του... Ε, δεν είναι εδώ η κυρία Κέπελ, όχι, επομένως ε, έχουν ε, μιλήσει όλοι όσοι είχαν εγγραφεί. Κύριε Πρόεδρε Μπούζεκ, ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε τις διαδικασίες έτσι ώστε να φτάσουμε στην πληροφορία όπως αρχικά είχαμε συμφωνήσει. Είναι πολλή δουλειά ε, αυτή που μας περιμένει. Ευχαριστώ τις εισηγήτριες για όσα έκαναν μέχρι τώρα. Ευχαριστώ βεβαίως ε, και τους σκιώδεις. Από όσο γνωρίζω, ήδη κάποιες συμβαστικές τροπολογίες είναι έτοιμες, όχι όλες. Έχετε κάνει φανταστική δουλειά. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι στην Επιτροπή Ήτρε είχαμε και μια έκθεση που ψηφίσαμε σήμερα για την Ενεργειακή Ένωση. Η ψηφοφορία μας πήρε περίπου δύο ώρες, αλλά μια χαρά τα καταφέραμε. Είμαστε ευτυχείς με το αποτέλεσμα και πέρασε μάλιστα το κείμενο με μεγάλη πλειοψηφία και με πάρα πολλές 50-60 δεν θυμάμαι συμβαστικές τροπολογίες. Επομένως σας εύχομαι τα καλύτερα και ε, όπως είπε και η Δίκη, θα προχωρήσουμε τώρα στο δεύτερο γύρο της συζήτησης που είναι οι other speakers, άλλοι ομιλητές πλην των ε, εισηγητών, σκιωδών κτλ. Από την ΙΜΚΟ ο πρώτος ομιλητής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η έκθεση εν τέλει πιστεύω ότι θα έχει σημαντική πνοή γιατί αυτό που κάνουμε είναι ζωτικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας μην κρυβόμαστε πίσω το δαχτυλό μας. Ε, ο, ανταγωνισμός ε, είναι παγκόσμιος. Ε, η Ευρώπη απέναντι στις Ηνωμένε Πολιτείε, απέναντι στην Ασία κτλ. Και νομίζω ότι η Ευρώπη τα προηγούμενα χρόνια έχασε το ραντεβού με το ψηφιακό κόσμο. Ε, είναι πολύ λίγες οι συσκευές, ε, οι ψηφιακές οι οποίες κατασκευάζονται στην Ευρώπη και οι πλατφόρμες που αναφέραμε προηγουμένως επίσης δεν είναι ευρωπαϊκές. Η έκθεση πρέπει να είναι λοιπόν ε, αισιόδοξη αλλά θα πρέπει να εκφράζει και ισχυρή θέληση θα πρέπει να αναφέρεται σε όλα αυτά τα οποία ε, θα πρέπει να κάνει η Ευρώπη για να γίνει ψηφιακή ε, με επενδύσεις, ε, με χρήση ιδιωτικών κονδυλίων και χρηματοδοτήσεων κτλ. Αλλά το μοντέλο αυτό θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τους πάντες γιατί εδώ μιλάμε για ένα νέο πρότυπο, ένα νέο μοντέλο κοινωνικό. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το σύνολο σύνολο των Ευρωπαίων πολιτών ε, θα ε, ε, έχουν πρόσβαση σε αυτή αυτά τα νέα στοιχεία έτσι ώστε να μπορέσουν να γίνουν ε, πλήρεις ε, ε, πρωταγωνιστές αυτής της νέας αγοράς και βεβαίως θα πρέπει όλοι οι οικονομικοί πρωταγωνιστές, όλοι οι φορείς και οι συμμετέχοντες να έχουν τον απαραίτητο βαθμό προστασίας. Ε, σας διαβεβαιώ πάντως ότι εάν δεν καταφέρουμε να νομοθετήσουμε ελάχιστα τουλάχιστον αλλά συνεκτικά, σας βεβαιώ ότι θα ε, προκύψουν ε, εθνικές ή μάλλον περιφερειακές νομοθεσίες οι οποίες θα δημιουργήσουν πρόβλημα. Δέστε τι γίνεται με την ε, Uber όπου οι αποφάσεις ε, είναι διαφορετικές μεταξύ τους. Θα πρέπει να φτάσουμε σε έναν ελάχιστο βαθμό ε, συμφωνίας αν ε, θέλουμε πραγματικά να έχουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Σας θυμίζω ότι στην αρχή του ηλεκτρονικού εμπορίου η έλλειψη εμπιστοσύνη ήταν μεγάλη και πολλοί ήταν διστακτικοί να μπουν Πρόκειται εδώ για την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση η οποία ε, ταυτοχρόνως είναι και κοινωνική επανάσταση. Δεν πρέπει να τη χάσουμε την επανάσταση αυτή για τις δύο εισηγήτρες τώρα δεν ξέρω αν το κείμενο θα είναι μακροσκελές περισσότερο, λιγότερο ή με περισσότερες λιγότερες σελίδες οπωσδήποτε όμως θα πρέπει να είναι αρκετά λεπτομερέ, γιατί θα πρέπει να δούμε τους ε, εμπλεκόμενους ε, ε, φορείς ε, εάν είναι λεπτομερές αλλά συνεκτικό δεν ε, υπάρχει πρόβλημα το, το, το πρόβλημα θα είναι αν είναι λεπτομερές αλλά και ασύνδετο για να τελειώσω δύο λόγια για το συνάδελφο που μόλις μίλησε όσον αφορά τα χρυσοιατικά δέντρα. Άλλωστε φτάνει σιγά σιγά ο Δεκέμβριος. Εγώ δεν θέλω το, το δέντρο το χριστουγεννιάτικο να είναι μόνο πράσινο, είναι μονότονο αυτό. Θέλω να έχει ωραία διακόσμηση γιατί όσο άσχημο και κακότεχνο είναι ένα κακοστολισμένο δέντρο τόσο όμορφο είναι όταν είναι όμορφα στολισμένο. Ε, εμείς, ε, λέει ο Πρόεδρος, είχαμε προβλέψει για την κατηγορία των άλλων ομιλητών δύο λεπτά. Εσείς μιλήσετε πολύ περισσότερο, πρέπει να προσέχετε συνάδελφοι. Δύο λεπτά ο καθένας. Κυρία Μόντι. Την Ήτρε. Uh, ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ και τις συνεισηγήτριες και τους ε, σκιώτες εισηγητές για τόσο σκληρή δουλειά που έχουν κάνει. Τρία εις παρατηρήσεις έχω σε σχέση με προηγούμενα σχόλια. Ε, το στόχος μας ε, είναι να καλύψουμε τα κενά που εντοπίζονται. Ποια είναι αυτά. Ένα από αυτά είναι ότι είμαστε αντιμέτωποι με νέα οικονομικά μοντέλα. Είναι ζωτική σημασία να εκπροσωπήσουμε τους πολίτες ε, στη δουλειά που κάνουμε, στο πώς προσεγγίζουμε το θέμα. Καθολική κάλυψη με ευρυζωνική σύνδεση πρόσβαση σε ε, διαρκή εκπαίδευση και κατάρτιση και το φαινόμενο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Και επίσης να καλύψουμε οπωσδήποτε την πτυχή της απασχόλησης στην ψηφιακή ενιαία αγορά. Είναι ζωτικής ε, σημασίας ο αντίκτυπος για τα κοινωνικά ζητήματα και την απασχόληση πρέπει οπωσδήποτε να συνυπολογιστεί και είναι θεμελιώδου σημασία να ληφθεί ε, υπόψη. Madam, Σας ευχαριστούμε. από την Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τις ε, εισηγήτριες. Νομίζω ότι ο αυξημένος αριθμός ε, των τροπολογιών δείχνει την επιθυμία των ε, βουλευτών να εργαστούν πάνω στο θέμα αυτό, αλλά βεβαίως και το μεγάλο ενδιαφέρον και τη σημασία αυτής της έκθεσης. Θα ήθελα να υπογραμμίσω δύο-τρία και να επιμείνω σε αυτά τα οποία έχουν αποτελέσει αντικείμενο δικών μου τροπολογιών πιστεύω ότι μπορούμε να συμβάλλουμε πολύ ουσιαστικά ε, στην ε, ψηφιακή αγορά και την ενιαία αγορά. Αυτός είναι ένας πολύ σημαντικός στόχος που θα μας δώσει τη δυνατότητα βέβαια να ε, βελτιώσουμε την εσωτερική αγορά, να δώσουμε νέα εργαλεία στην αγορά αυτή. Η ενιαία ψηφιακή αγορά που θα πρέπει να είναι βεβαίως δίκαιη και ομοιογενής ε, θα δώσει μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα στην ε, βιομηχανία, θα δώσει όθηση ε, και στις νεοφυείς αλλά και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα προστατέψει πιο αποτελεσματικά τα δικαιώματα των καταναλωτών και θα υπεραμεινθεί μιας υγιούς πολιτικής ανταγωνισμού. Όσον αφορά τα θέματα που με απασχόλησαν, έχω υποβάλει κάποια ερωτήματα ε, και κάποια ζητήματα. Πρώτον, να ε, ε, ε, λάβουμε υπόψη μας και να προωθήσουμε όλα τα στοιχεία τα οποία μας έρχονται από τη συμμετοχική οικονομία που θα λαμβάνουν βεβαίως υπόψη το, την ανάγκη να, μην, να προστατέψουμε τους τομείς και όχι να τους κυρώσουμε. Ένα επίσης μια ίδια αντιμετώπιση όλων όσον αφορά τις ε, φορολογικές απαιτήσει και όσον αφορά την καταβολή των φόρων. Ένα άλλο θέμα είναι ε, το θέμα της κατάργησης ε, του γεωαποκλεισμού, του geo-blocking όλες αυτές οι μορφές οι οποίες ε, ε, ε, μεταχειρίζονται με διακριτικό τρόπο, με διαφορετικό τρόπο τους καταναλωτές δεν μπορεί να μας βρει σύμφωνους. Ένα άλλο θέμα είναι η ανάγκη επένδυσης μεγαλύτερων, περισσότερων πόρων για την ασφάλεια των δικτύων. Έχουμε διαπιστώσει ότι συχνά οι καταναλωτές έχουν προδοθεί από ανασφαλή δίκτυα και επομένως έχει αρθεί η εμπιστοσύνη τους στο υφιστάμενο σύστημα προστασίας των των δικτύων. Θα πρέπει μέσω επενδύσεων λοιπόν να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Τέλος, μεγάλη επένδυση στο σύστημα διακυβέρνησης έτσι ώστε η ε, εθνική διοίκηση αλλά και η ευρωπαϊκή ευελπιστό διοίκηση θα γίνει πιο φιλική προς τον τελικό χρήστη που είναι ο ε, Ευρωπαίος καταναλωτής. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λοιπόν. Υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο όνομα. Ρούζα, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Long name, but short intervention. Μικρό το όνομα, μικρή και η παρέμβασή μου, λοιπόν. Κοιτάξτε, εγώ τη στιγμή που καταφέραμε να βρούμε μία λύση για τις χρεώσεις της περιαγωγής Αναμένω να βρούμε και μία λύση για τις υπηρεσίες τις ταχυδρομικές τη στιγμή που αναπτύσσεται τόσο γρήγορα το ηλεκτρονικό εμπόριο γιατί είναι κάτι που οι πολίτες θέλουν να λύσουμε. Έχουμε κάποιες συμβαστικές προτάσεις και εγώ έχω υποβάλει συμβαστικές τροπολογίες και θέλω να τις πάρουν σοβαρά οι εισηγητές. Αλλά δεν αρκούν αυτά. Πρέπει να λυθεί το ζήτημα. Ε, τι αν υπάρχουν εσωτερικά σύνορα στην ε, ενιαία αγορά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κρίλ. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα την εισηγήτρια. Πάρα πολύ καλή δουλειά. Επίσης υπάρχει ένα σημείο όμως στην έκθεση που ζητάει ε, μια Ευρωπαϊκή Ρυθμιστική Αρχή ε, για τις τηλεπικοινωνίες. Λάθος. Υπάρχει η BERIC και υπάρχει ακριβώς ε, όπως είπαμε η BERIC, αυτή η οποία είναι δηλαδή μια συνεργασία των εθνικών ρυθμιστικών αρχών η οποία λειτουργεί μια χαρά. Και δεν πρέπει τώρα μέσα στη μέση να αλλάζουμε την ε, κατάσταση για τους κανόνες του παιχνιδιού απλά θα πρέπει να παραμείνουμε στη συνεννόηση που υπάρχει δεν νομίζω να χρειάζεται εδώ πέρα Ευρωπαϊκή Ρυθμιστική Αρχή και νομίζω πως συμφωνούμε με τους συναδέλφους Ευχαριστώ Ο κύριος Ντάλτον από την ΕΜΚΟ Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ για την καλή συνεργασία. Ευχαριστώ τι συγκίτρε και του κοιόδε. Έχω καταθέσει διάφορε τροπολογίε για διάφορα ζητήματα. Θα σχολιάσω όμω μόνο κάποια από αυτά. Πρώτον, ο χειρό Ευρώπη, είτε μιλάμε για την ασφάλεια στο υπολογιστικό νεφο ή για το περιεχόμενο, πρέπει οπωσδήποτε να μην αποκόψουμε την Ευρώπη από τον υπόλοιπο κόσμο, γιατί η παγκοσμιοποίηση μεγενθύνεται κάθε μέρα. Εμεί δεν μπορούμε να είμαστε σε, ε, απομονωμένοι σε ένα ψηφιακό νησί. Θα τιμωρήσουμε του καταναλωτέ. Ε, το άτομο πρέπει να είναι στην καρδιά όλων όσων κάνουμε. Θα πρέπει επίση ε, να ενισχύσουμε την ισχύ που έχουν οι καταναλωτές και να μην μπαίνουν μέσα στη μέση οι, πολιτές, οι πολιτικές. Συγγνώμη. Επίσης χρειαζόμαστε φορητότητα των δικαιωμάτων ε, και οι φραγμοί που υπάρχουν, οι αποκλεισμοί που υπάρχουν ε, εμποδίζουν αυτήν την κινητικότητα και αυτό είναι επιζήμιο για την πνευματική δημιουργία. Θα ήθελα επίσης να απευθυνθώ στους αντιπρόεδρους. Αναμεταδίδεται στο διαδίκτυο ε, η συνεδρίαση. Υπάρχει γεωαποκλεισμό. Φαντάζομαι ότι αναμεταδίδεται στον κόσμο όλα αλλά πρέπει να το ε, διευκρινίσουμε αυτό. Ε, γιατί, διότι υπάρχει ο αποκλεισμό και εσείς προσθέτετε αυτά που θέλετε να αποκλείσετε. Είναι μια default λειτουργία. Θα ήθελα τώρα να επιμείνω ε, σε σχέση με τις υπηρεσίες που πρέπει να υπάρχουν σε όλες τις χώρες, όπως το Uber. Πώς γίνεται, ας πούμε, αλλού να υπάρχει, αλλού να μην υπάρχει. Τι ενιαία αγορά είναι αυτή και το ένα πολύ σημαντικό με τις ψηφιακές οικονομίες είναι ότι υπάρχει μεγάλη αποτελεσματικότητα διότι η προσφορά ε, ε, αντιστοιχεί στη ζήτηση και νομίζω ότι πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό. για τις συνεργατικές οικονομίες θα πρέπει να ε, ε, επιταχύνουμε την ίδρυση μιας επιχείρησης μέσα σε μία μέρα θα πρέπει να είναι δυνατόν οτιδήποτε ε, μεγαλύτερο θα, μας, θα έχει ως αποτέλεσμα να υστερούμε σε σχέση με τις ΙΠΑ. Λοιπόν, η ενιαία αγορά θα πρέπει να είναι στην υπηρεσία κυρίως των επιχειρήσεων και των καταναλωτών. Απάντηση της Βίκη Φόρντ δεν υπάρχει για αποκλεισμό. Είναι διαθέσιμη παγκοσμίω η αναμετάδοση. Ευχαριστούμε κυρία Ροζιέρο.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 Όλα αυτά τα μεγάλα ζητήματα ε, τα οποία σχετίζονται με την ψηφιακή αγορά είναι πάρα πολλά και πολύ σημαντικά για να μην τα λάβουμε υπόψη μας. Ωστόσο, οι στόχοι μας δεν θα επιτευχθούν εάν δεν επιτύχουμε πρώτα πραγματική εναρμόνιση και όχι μονάχα εναρμόνιση στην πρόσβαση στις υπηρεσίες, αλλά ε, μια εναρμόνιση η οποία θα αφορά το σύνολο της ε, δραστηριότητας που θα αφορά τις τα κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων πούμε ε, γιατί τώρα ε, συχνά ε, στην συμμετοχική οικονομία απλά μας παρουσιάζεται ένα οικονομικό μοντέλο όπου καταπατώνται και παραβιάζονται τα κοινωνικά και εργατικά εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων. Επομένως τα, οι, οι κοινωνικοί προβληματισμοί, οι περιβαλλοντικοί προβληματισμοί είναι για μας πάρα πολύ σημαντικά. Ε, τώρα, ε, ένα, οι συγγραφείς, οι ε, δημιουργοί που είναι μια ειδική κατηγορία εργαζομένων, ξέρουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις έχουμε πολλές μεγάλες εταιρείες οι οποίες δεν είναι ευρωπαϊκές και οι οποίες καταπατούν κατάφορα τα δικαιώματα των δημιουργών. Τέλος, για να αποφύγουμε αυτούς τους ε, μηχανισμούς ε, ε, των μη, της αντιδιαστολής των μη εναρμονισμένων νομοθεσιών, θα πρέπει εμείς να απαντήσουμε με μια ισχυρά ενοποιημένη, ομοιογενοποιημένη νομοθεσία, η οποία δεν θα δίνει κανένα περιθώριο, δεν θα αφήνει κανένα περιθώριο για παραβίαση κοινωνικών εργασιακών δικαιωμάτων δικαιωμάτων. Έχουμε, τα έχουμε συζητήσει αυτά και στην Επιτροπή μας εδώ και ένα χρόνο τα συζητούμε ε, και γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι πραγματικά μπορούμε να δημιουργήσουμε μια σωστή ψηφιακή αγορά. Thank you very much, Madame. Madame Griffin is the next speaker. Thank you, Chair, and thank you to the... Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Γκρίφη. Ευχαριστώ τις συγγήτριες. Ε, θα ήθελα να στηρίξω ε, και αυτό που είπαν και άλλοι ομιλητέ σχετικά με την ανάγκη προστασίας ε, των κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων ε, των πολιτών. Θέλουμε πρόσβαση επίσης και των πιο ευάλωτων πολιτών στην την ε, ε, ψηφιακή οικονομία. Κατά 40% έπεσε στην Κάμπρια, στη δική μου δηλαδή εκλογική περιφέρεια, η χρήση της 4G. Ε, αυτό δεν είναι δυνατόν να το δεχτούμε. Επίσης θέλουμε εργασία, θέσεις εργασίας, οι οποίες θα δίνουν πραγματικά προστιθέμενη αξία. Mr. Blanco Ευχαριστώ πολύ. Ναι, πρέπει να παρέμβω στην Επιτροπή ε, Αλληλείας για ένα θέμα για το οποίο είμαι εισηγητής, γι' αυτό βιάζομαι. Ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τις εισηγήτριες. Ε, αν δεν το έχετε καταλάβει, ε, πλέον πρέπει, πλέον έρονται τα όρια ανάμεσα στο φυσικό και το ψηφιακό κόσμο και τώρα είναι η στιγμή που πρέπει να κάνουμε πιο σημαντική και αποτελεσματική νομοθέτηση θα πρέπει οπωσδήποτε ε, να ε, βελτιώσουμε, να διορθώσουμε ε, τα, τα πλαίσια τα οποία τα νομοθετικά τα οποία θα διορθώσουν τις τρευλώσεις. Το είδαμε με τα απατηλά τεστ της, και το πειραγμένο λογισμικό της Volkswagen. Επίσης πρέπει να μάθουμε από τα λάθη του παρελθόντος, ε, να αποφύγουμε λάθη προηγούμενων ενώσεων όπως ε, της νομισματικής ε, και να δώσουμε όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία θα επιτρέπουν την ισομερή, ισοδίκαιη πρόσβαση όλων των πολιτών. Επίσης θα πρέπει με εναρμονισμένους κανόνες να προχωρήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο έτσι ώστε κανείς να μην θεωρεί ότι μόνος του μπορεί να αντιμετωπίσει τις προϋποθέσεις και τις ε, προκλήσεις ε, της ψηφιακής ε, κοινωνίας. Τα κύρια στοιχεία μας θα πρέπει να αναφέρονται στην προστασία των καταναλωτών, στην ασφάλεια του δικτύου, στην προστασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και όλων όσοι λειτουργούν στα πλαίσια του ψηφιακού κόσμου, κυρίως με αυτούς που ασχολούνται με την ε, με την έρευνα και την καινοτομία ε, αλλά κατά την άποψή μου όπως όλα όσα σχετίζονται με την βελτίωση και εξυγχρονισμό ε, του πλαισίου της προστασίας της, ε, των πνευματικών δικαιωμάτων ε, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και θα πρέπει ταυτοχρόνως να δούμε την νομική διευθέτηση των πλατφορμών, των ενδιαμέσων κλπ. Είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι η κοινή μας εργασία θα δώσει κατευθυντήριες γραμμές προς την Κομισιόν έτσι ώστε να μπορέσουμε σε αυτή σε αυτό το κοινοβούλιο να παίξουμε σημαντικό ρόλο τους μήνες που έρχονται. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους εκπροσώπους ε, των δύο επιτροπών. Να σας υπενθυμίσω, συνάδελφοι, πως έχουμε πολλές επιτροπές. Η ΙΜΚΟ και η ΙΤΡΕ είναι κατά κύριο λόγο με βάση το άρθρο 54 και μετά έχουμε όπως είπαμε τις επιτροπές απασχόλησης Γιούρι και ΛΥΜΠΕ και έχουμε και απλές γνωμοδοτήσεις ε, Επιτροπή ΕΚΟ και Μεταφορών και Αλίες. Εννέα επιτροπές συνολικά. Αρκετές. Ο κύριος Νίλσον λοιπόν από την ΙΜΚΟ κατόπιν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η ψηφιοποίηση δημιουργεί νέες μεγάλες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και για τους καταναλωτές. Εγώ θεωρώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να περάσει το εξή μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν θα πρέπει να προωθήσουμε άκρητα ε, τα νέα επιχειρησιακά μοντέλα, τα ευφυή επιχειρησιακά μοντέλα. Θα πρέπει να προστατεύσουμε και τους καταναλωτές ε, για την ε, ψηφιοποίηση. Υπάρχουν και σοβαρά θέματα, όπως παραδείγματος χαρή, οι φορολογικές αρχές που εποπτεύουν την κατάσταση και εισπράττουν τα φορολογικά έσοδα. Μόνο έτσι μπορεί να λειτουργήσει ένα κράτος πρόνοιας και θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα σε τέτοιες υπηρεσίες. Θα πρέπει επίσης συνειδητοποιήσουμε ότι ε, έρχονται σε εμά ε, μικρές επιχειρήσεις ε, και τους λέμε τι, ότι μπορεί να τους βοηθήσει ο νέος ψηφιακός κόσμος γιατί έτσι μπορούν να μην πληρώνουν του φόρου ή να μην έχουν να πληρώνουν τόσο υψηλές κοινωνικέ εισφορές. Υπάρχουν σοβαρές παρανοήσεις και νομίζω ότι μέσα στην εγγονότηση του Κοινοβουλίου πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε ξεχωριστό κεφάλαιο για τα κοινωνικά ζητήματα. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Σύνφελ από την ε, Επιτροπή ε, ΙΜΚΟΜ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η ψηφιακή αγορά δεν είναι ούτε ευρωπαϊκή ούτε αμερικανική. Είναι παγκόσμια παρά το ότι ε, εμείς απλοποιούμε τα πράγματα. Υπάρχουν λοιπόν δύο σχολές σκέψης. Η μία είναι το να προστατεύσουμε την αγορά, να σκεφτόμαστε τα δικαιώματα των καταναλωτών και των χρηστών, η Αμερικανική σχολή. Και... Μετά έχουμε την ευρωπαϊκή σκοπιά, να προστατεύουμε τους χρήστες και τα λοιπά. Αλλά αν δούμε την ψηφιακή αγορά βλέπουμε πως η Ευρώπη μένει πίσω. Πρέπει να θυμόμαστε πως η υπερβολική ρύθμιση της αγοράς μπορεί να καταστήσει την Ευρώπη μη ανταγωνιστική όχι μόνο απέναντι στη ΣΥΠΑ αλλά και σε άλλα μέρη του κόσμου γιατί και οι άλλες περιοχές του κόσμου έχουν βεβαίω ε, τις ευκαιρίες τους και δεν θα μας περιμένουν. Ο μόνος τρόπος που μπορούν να ανταγωνιστούν τις ΕΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ακριβώς μέσω του ψηφιακού φάσματος. Αλλιώς, αν δεν το καταλάβουμε αυτό, θα συνεχίσουμε εμείς εδώ πέρα να εγκρίνουμε νομοθεσία κτλ. που δεν θα έχουν σχέση με τον πραγματικό κόσμο. Και ε, βλέπουμε πως οι νέες εταιρείες ξεκινάνε στη ΣΥΠΑ. Δεν ιδρύονται στην Ευρώπη. Και αυτές που ιδρύθηκαν στην Ευρώπη πηγαίνουν στην Αμερική. Γιατί είναι καλύτερο το επιχειρηματικό περιβάλλον. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε πώς θα δημιουργήσουμε μια αγορά φιλική στις επιχειρήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Γκαλπέλτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω πως είναι, ένα, είναι πάρα πολύ σημαντική και χρήσιμη αυτή η συζήτηση. Είναι η δεύτερη φορά που συζητάμε αυτό το θέμα, αλλά πρέπει να θυμόμαστε ποιοι θα ωφεληθούν οι ευρωπαϊκές εταιρείες και άρα οι ευρωπαίοι πολίτες αλλά για να κάνουμε κάτι τέτοιο πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτές τις ευκαιρίες θα ήθελα τώρα να εστιαστώ στην προστασία δεδομένων γιατί τα δεδομένα είναι και ευκαιρία και κίνδυνος. Για τις ευρωπαϊκές εταιρείες η διαχείριση των δεδομένων κρίνει την ανταγωνιστικότητά τους. Σίγουρα όλοι συμφωνούμε πως η πληροφορία είναι ισχύς. Τα δεδομένα δηλαδή. Προσπαθούμε, προσπαθούν οι ευρωπαϊκές εταιρείε να είναι ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο και δεν τα πάμε και πολύ καλά. Λοιπόν, για να μπορέσουμε να κινηθούμε καλύτερα στον παγκόσμιο ανταγωνισμό, πρέπει να αλλάξουν οι κανόνες προστασίας δεδομένων, να είμαστε πολύ πιο ρεαλιστικοί. Και εγώ θα ήθελα η έκθεση αυτή να συνεισφέρει κάπως όπως είπε και ο προηγούμενος ομιλητής στο να γίνουν οι ευρωπαϊκές εταιρείες πιο ανταγωνιστικές και να φτάσουν τις αμερικανικές εταιρείες γιατί θέμε πιο ανταγωνιστικές εταιρείες ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνουμε κάτι ουσιαστικό όχι άλλο ένα χαρτί Ευχαριστώ κύριο Σουάμπ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Παρακολούθησα προσεκτικά τη συζήτηση. Είναι νομίζω μια καλή βάση το σχέδιο έκθεσης της συναδέλφου και τις 1200 ε, τροπολογίες ε, που είδα. Πρέπει να δούμε δύο πράγματα εδώ πέρα, να δούμε το ρόλο που θα παίξουν στην έκθεση. Έχουμε το τι γίνεται με τους εργαζόμενους και τα συμφέροντα των εργαζομένων που θα επομιστούν ε, και βλέπουν με ανησυχία το θέμα της αλλαγής της αγοράς εργασίας και βεβαίω εδώ πέρα η έκθεση αυτή είναι μια κάποια απάντηση του Κοινοβουλίου στην Κομισιόν και το άλλο θέμα είναι το θέμα της φορολογικής πολιτικής που παίζει διαφορετικό ρόλο στον ψηφιακό κόσμο, αλλά επί της αρχής θεωρώ πως το βασικό μήνυμα της έκθεσης πρέπει να είναι ότι εμείς ως Κοινοβούλιο θέλουμε ίσους όρους ανταγωνισμού ανεξαρτήτως το που βρίσκεται κάποιος στην Ευρώπη και οι κανόνες να μεταφέρονται στον ψηφιακό κόσμο έτσι ώστε μια εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται με τον παραδοσιακό τρόπο να μην έχει μειονέκτημα. Πρέπει λοιπόν να δούμε το ερώτημα ποιους παλιούς κανόνες πρέπει να επεξεργαστούμε έτσι ώστε να είναι ίση η όρη του ανταγωνισμού ανεξαρτήτως ε, του πιο ποιον διάβλο επιλέγει μια εταιρεία. Εδώ πέρα λοιπόν πρέπει να τοποθετηθούμε σαφώς, γι' αυτό θα ήθελα να ζητήσω και του αδελφού την όσο δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Στήλερ. Ναι. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τις συνεισηγήτριες. Ε, πολλά υπόθηκαν ε, σε σχέση με το πόσο σημαντική είναι η ψηφιακή αγορά. Εγώ ήθελα να σχολιάσω μόνο κάτι που ακούσαμε για τα δεδομένα. Στο ψηφιακό σύμπαν ε, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι μέχρι το 2020 θα έχουμε 44-3 σε όλα αυτά τα δεδομένα έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία δύο χρόνια και υπάρχουν ε, χιλιάδες επιστημονικά έρθρα για αυτά και επειδή θα μας απασχολεί στα πλαίσια της έκθεσης θα πρέπει να το συζητήσουμε. Ε, η Φιλανδή συνάδελφος ε, το ανέφερε διότι βασικοί ερευνητές μας μιλάνε για την σημασία της έρευνας σε σχέση με αυτές τις εκατοντάδες ε, χιλιάδες, ε, εκατοντάδες χιλιάδες τομείς όπου θα έχουμε τόσο πολλά δεδομένα. Ε, υπάρχει και το θέμα της έρευνας, του data mining των δεδομένων. Νομίζω ότι αυτό δεν ακούστηκε καθόλου συζήτηση. Ένα παράδειγμα, μια φαρμακευτική εταιρεία, παραδείγματο χάρη, σε 18 μήνε εξετάζει 500.000 σε διπλώματα ευρεσιτεχνία. Ε, αν δείτε ποιο είναι το δυναμικό, ε, πόσο χρόνο και χρήμα μπορούμε να εξοικονομήσουμε αν είμαστε πιο καινοτόμοι για την μεταχείριση των δεδομένων, ε, θα καταλάβετε πόσο μεγάλη σημασία έχει αυτό στα πλαίσια τη ενιαίας ψηφιακή αγορά, Ευχαριστώ και προσπάθησα να μην ξεπεράσω και το χρόνο μου μου. Σας ευχαριστούμε κυρία μου. Θέλαμε τώρα να ακούσουμε την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. έχετε συντάξει την ανακοίνωση. Ο κ. Ζεράρτε γράφει αρμόδιος για την ψηφιακή ενιαία αγορά, για το συντονισμό της ψηφιακή ενιαίας αγοράς στη ΔΕΛΤΑ κονέκτε, θα πάρει το λόγο. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Αγαπητά μέλη της Επιτροπής, ε, θα μιλήσουμε δύο ε, για αυτό το θέμα και από τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ε, η συνάδελφος εδώ δίπλα μου θα ακολουθήσει. Λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι ε, είναι πολύ σημαντικό γιατί εδώ αναφέρω τα βασικά ζητήματα και επίσης ε, συνειδητοποιείται πόσο επίγον είναι το ζήτημα ότι γρήγορα θα πρέπει να λάβουμε ε, τις δικές σας θέσεις για να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε και να ολοκληρώσουμε αυτή την ενιαία ψηφιακή αγορά. Ως προς τη μεθοδολογία, διότι όντω υπάρχει κατακαιρματισμός στην ενιαία αγορά, θα πρέπει να τεθεί το ζήτημα πρώτα απ' όλα Πώς συνέβη αυτό. Ε, αν κοιτάξουμε ε, τις ε, νομοτεχνικές εργασίες ε, των τελευταίων ετών θα διαπιστώσουμε ότι υπήρξε μια ελάχιστη εναρμόνιση χάρη στην οποία μπόρεσαν κάποια κράτη-μέλη να ε, προοδεύσουν. Όμως ο στόχος θα πρέπει να είναι ένας ενίος κανός και όχι 28 διαφορετικοί που ε, και δεν θέλουμε 28 συν ένα κανόνα, 29, θέλουμε έναν ενίο κανόνα. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας, να έχουμε ίσους ε, όρους ε, ανταγωνισμού, το ανταγωνισμό και έτσι οι καταναλωτές, επιχειρήσεις και ιδιώτες θα έχουν αυξημένη εμπιστοσύνη και θα μπορέσουν ευκολότερα να κινηθούν σε άλλες χώρες για τις δύο συνοριακές συναλλαγές. Μια startup, παραδείγματο χάρη, ξέρει ότι δεν πρέπει να αρχίσει 28 διαφορετικές φορές για να δραστηριοποιείται σε όλη την Ευρώπη. για μια μεγάλη εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει τα μεγάλα δεδομένα, τα big data, Τη της οικονομίας σε κλίμακας μέσα στο υπολογιστικό νέφος μόνο εάν νιώθει ε, Πιστοσύνη για το γεωαποκλεισμό. Εμείς έχουμε εργαστεί σκληρά γι' αυτό, διότι υπάρχει και το θέμα του γεωαποκλεισμού περιεχομένου που προστατεύεται ε, ως προς τα πνευματικά δικαιώματα. Αυτή είναι η διαφορετική πρόταση. Τις επόμενες, ε, τους επόμενους μήνες θα καταθέσουμε πρόταση για τη φορητότητα των δικαιωμάτων. Αυτό είναι το ένα θέμα. Και το άλλο θέμα είναι ο γεωαποκλεισμός για το περιεχόμενο που δεν ε, προστατεύεται ως προς τα πνευματικά δικαιώματα. Θα ακολουθήσει διαφορετική πρόταση για της πλατφόρμας. Ενδιαφέρον θέμα Όμως, ακόμη σημαντικότερο είναι ποιο είναι το πρόβλημα που προσπαθούμε να λύσουμε. Υπάρχει πρόβλημα που πρέπει να λύσουμε, τότε ε, ε, να αποφασίσουμε αν η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και το, ο καλύτερος ε, τόπος και τρόπος για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα, εάν υπάρχει, διότι ασχολούμαστε με τον ορισμό και μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε ότι επειδή είναι τόσο διαφορετική, το δεν έχει νόημα ένα ορισμό ε, για τι πλατφόρμε. Ε, ε, Πολλέ πτυχέ καλύπτονται από την κείμενη νομοθεσία. Ποιο είναι ο ρόλο τη πλατφόρμα για την αναθεώρηση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών για τη, τη γραμμικότητα, η μη γραμμικότητα, για τα πνευματικά δικαιώματα, για τις οπτικοακουστικές υπηρεσίε, Σε αυτού του Όμω έχει σημασία ορισμός, αν θέλετε, τη πλατφόρμα, αλλά έχει διαφορετικές εκφάνσεις. Ε, τώρα θα ακούσουμε τη συνάδελφό μου, η κυρία Μάρεν Γκρούμπεν, ε, γιατί υπεύθυνη στη γάμα Δέλτα Growth ανάπτυξη για την ψηφιοποίηση της ενιαίας αγοράς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάποια σχόλια ήθελα να κάνω σε κάποια πράγματα που είπαν αρκετοί ομιλητέ. Το ένα αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό της βιομηχανία. Κάποιοι θεωρούσατε πως δεν το είχαμε τονίσει αρκετά. Ο Αντιπρόεδρος Κατάινεν πρόσφατα είπε πως σκοπεύει να κάνει μια ομάδα εντός της, ομα... εντός Κομισιόν για να δει ακριβώς ε, τι γίνεται στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της βιομηχανίας. Και βεβαίως εδώ πέρα μιλάω για τις επενδύσεις που έρχονται από διάφορα μέσα, τη δουλειά που συνεχίζεται στην οικονομία των δεδομένων, το ίντερνετ των πραγμάτων, ζητήματα τυποποίησης και διαλειτουργικότητας και βεβαίως η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων. Σκοπεύουμε λοιπόν να δούμε πιο στενά τα πακέτα αυτά και να βελτιωθεί η αφήγηση σε σχέση με τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Το άλλο αφορά την δηλωτική οικονομία στην η οποία βεβαίως απασχολεί μεγάλο κομμάτι της ανακοίνωσής μας. Υπήρχε ένα κεφάλαιο που είχε ήδη ανακοινωθεί. Τι σκοπεύουμε λοιπόν να κάνουμε στα μέσα του επόμενου έτους να έχουμε εμένα μια ευρωπαϊκή ατζέντα για το θέμα αυτό που θα μας οδηγήσει στην εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων και θα δημιουργήσει ένα πλαίσιο παρακολούθησης ε, για να δούμε, να δούμε τι γίνεται στην συνεργατική οικονομία. Γιατί βεβαίως θεωρούμε πως ε, η δυνατότητα που υπάρχει οι δυνατότητες που υπάρχουν είναι πάρα πολύ μεγάλες καινοτόμα ζητήματα που αναπτύσσονται εκεί και οι δυνατότητες ε, που προσφέρουν για επανένταξη στην αγορά εργασίας ε, το πώς ε, κινητοποιεί την επιχειρηματικότητα όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα αλλά ταυτόχρονα όπως είπατε υπάρχουν και προκλήσεις και απειλές πολλοί έρχονται σε εμά και παραπονιούνται για το ότι δεν υπάρχει νομική σαφήνεια δεν ξέρουν πώς θα εφαρμοστούν οι κανόνες μιλάνε για κανόνες δυσανάλογους και επίσης παραπονιούνται για τον κατακερματισμό του ρυθμιστικού πλαισίου στα κράτη-μέλη. Προφανώς οι παραδοσιακές εταιρείε παραπονιούνται για την έλλειψη ίσου ανταγωνισμού και τα κράτη-μέλη ανησυχούν για φόρους, ε, εισφορές ε, κτλ. Τα γνωρίζουμε όλα αυτά. Θα συνεχίσουμε λοιπόν όπως είπαμε με τα διαφορά εργαστήρια. Θα μιλήσουμε με τους επιχειρηματίες και με βάση αυτά και βεβαίω τη δική σας συνεισφορά ελπίζουμε να καταλήξουμε σε κάποιες κοινέ λύσεις έτσι ώστε να υπάρχει νομική βεβαιότητα για τους επιχειρηματίες να υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο θετικό για την ανάπτυξη και τις δουλειές να μπορέσουν οι κατανολτές να αποφεληθούν και τέλος να αποφύγουμε τον περαιτέρω κατακαιρματισμό της ενιαίας αγοράς γιατί εάν γίνει κάτι τέτοιο τότε όλες αυτές οι πολλοεποσχόμενες εταιρείε δεν θα μπορέσουν ποτέ να ανέβουν κατηγορία σας ευχαριστώ περνάμε ξανά στους ηγητές κυρία Γκέπχαρτ ευχαριστώ κύριε πρόεδρε πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και ευχαριστώ όλους τους ε, συναδέλφους Νομίζω λοιπόν πως ε, κάτι θα μπορέσουμε να κάνουμε. Πρώτα απ' όλα να πω πως συμφωνώ με τις διαπιστώσεις ε, του κυρίου Μπούζεκ και της κυρίας Φόρντ. Δεν πρέπει να αναβάλουμε καθόλου την ε, υπόθεση. Πρέπει αντιθέτως να υπάρξει κάποια αντίδραση του Κοινοβουλίου. Γι' αυτό ναι, ακροάσεις ευχαρίστως αλλά όχι αναβολή της ψηφοφορίας. Σας παρακαλώ. Θα πρέπει να γίνουν και άλλες εκθέσεις από ό,τι φαίνεται στο θέμα αυτό. Οπότε πρέπει να ξεκινήσουμε. Για τον κύριο Ζιβέν να πω πως προσπαθούμε να καταλήξουμε σε κάποιες συμβιβαστικές προτάσεις το συντομότερο δυνατόν. Πιέζει ο χρόνος και δεν είναι απλό το πράγμα αυτό, δηλαδή να συμφωνήσει, να συμφωνήσουμε με τον κύριο Κάλλας. Προσπαθούμε λοιπόν να εργαστούμε όσο δυνατόν πιο γρήγορα γιατί γνωρίζουμε πως ε, εντάξει, η ιδανική εργασία γίνεται με άφθονο χρόνο. Προσπαθούμε λοιπόν, σας το υπόσχομαι, χωρίς να θέλω να υπόσχομαι πράγματα που δεν μπορώ να κάνω. Λοιπόν, κύριε Τσούλο, το θέμα μας δεν είναι εδώ πέρα τώρα να ικανοποιήσουμε τους πάντες, δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Προσπαθούμε να έχουμε ε, ένα ενιαίο όραμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο οποίο θα συμφωνήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι βουλευτές χωρίς να νερώσουμε τα πράγματα. Γι' αυτό απορρίπτω αυτό το οποίο είπατε ότι θα γίνεται forum shopping και θα διαλέγει ο καθένας που θα για το περιεχόμενο. Κάτι ε, πρόσεξα στη συζήτηση. Όλοι θα είναι μια θετική προσέγγιση. και συμφωνούμε όλοι σε αυτό αλλά συχνά έχω την εντύπωση πως παρουσιάζουμε τα πράγματα λίγο μαύρα δεν είναι τόσο άσχημη η οικονομία μας όσο είπαν μερικοί συνάδελφοι να σας παρακαλέσω να μην κάνετε αυτό που κάνουν μερικοί Μην δημιουργήσουμε δηλαδή την εντύπωση πως ε, δεν αξίζει να μείνει ένας νέος επιχειρηματίας στην Ευρώπη και καλά θα κάνει να φύγει. καλό να είστε λίγο προσεκτικοί. Γιατί βεβαίω θέλουμε να ε, ε, εκμεταλλευτούμε αυτή τη δημιουργικότητα. Δεν μπορεί να πάνε όλοι στην Silicon Valley. Οπότε δεν είναι δυνατόν να παρουσιάζουμε τα πράγματα πιο μαύρα από όσο είναι. Τώρα να έρθω στο περίφημο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Πλησιάζουν κάπως και τα Χριστούγεννα και το συζητάμε. Είναι συζητήσιμο το εάν το χριστουγεννιάτικο δέντρο ή όχι, αλλά εάν έχουμε χριστουγεννιάτικο δέντρο θα πρέπει να είναι λογικά ωραίο και στολισμένο και χρωμάτιστο για να είναι όλοι χαρούμενοι Οπότε πρέπει να υπάρχει μια συνέπεια και να μην γίνεται χαμός γιατί θα είναι άσχημο τότε το δέντρο. Λοιπόν, να πρέπει επίσης και το είπε ο κύριος Ντεγκράφ να δούμε το ποια προβλήματα πρέπει να λυθούν και πώς. Αυτά είναι τα ερωτήματα πρέπει να θέσουμε και βεβαίως πρέπει να προσέξουμε να μην έχουμε ένα μοσαϊκό μετά με 28 διαφορετικές ρυθμίσεις γιατί δεν κάναμε τίποτα στο ευρωπαϊκό επίπεδο και μετά να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε την κατάσταση που θα έχει δημιουργηθεί ειδικά το μιλάμε για τον γεωαποκλεισμό για τις πλατφόρμες για οτιδήποτε αφορά και μπορεί να ρυθμιστεί στην εσωτερική αγορά. Και πέρα πρέπει να το σκεφτούμε αν θέλουμε να το αφήσουμε στο εθνικό επίπεδο ή αν πρέπει να το ρυθμίσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και κάτι άλλο θα ήθελα να ξεκαθαρίσω εδώ. Κύριε Ντεγκράφ, μην προσπαθείτε να βρείτε έναν ορισμό για την πλατφόρμα. Θα αποτύχετε. Γιατί οι πλατφόρμες που προσφέρονται και πολλαπλασιάζονται συνεχώς και είναι τόσο διαφορετικές ώστε δεν θα βρείτε ορισμό. Μην χάνετε λοιπόν το χρόνο σας. Άντε δούμε που υπάρχουν προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Και έτσι βλέπουμε πως υπάρχουν διαφορετικά προβλήματα σε διαφορετικές πλατφόρμες. Σε πλατφόρμα του e-commerce υπάρχει το θέμα του γεωαποκλεισμού. Στην ε, συμμετοχική οικονομία υπάρχει το πρόβλημα των ψευδοαυτοαπασχολούμενων και τα σχετικά κοινωνικά προβλήματα. Στις μηχανές αναζήτησης έχουμε το πρόβλημα της ε, μονοπωλιακής θέσης κάποιων. Τελείως διαφορετικά δηλαδή προβλήματα σε διαφορετικούς τομείς. Και αυτή πρέπει να είναι και η προσέγγιση μας. Και εδώ τελειώνω. Παρά το ότι είχα και άλλα να πω. Uh, thank Σας ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Καλιάκάλα. Παρακαλώ. Και ευχαριστώ όλους όσοι πήραν το λόγο. Με χαρά διαπιστώνω ότι ε, οι περισσότεροι θεωρούν ότι αυτή η αισιόδοξη ε, λογική της έκθεσης πρέπει να παραμείνει. Το ζήτημα είναι ε, η, η συμμετοχική οικονομία ή ε, οι, οι πολίτες εάν εφαρμόσουμε με ίδιο τρόπο όλους τους κανόνες γιατί όλοι λένε ότι τα νέα εργαλεία δίνουν μεγαλύτερη ε, δύναμη στους καταναλωτές και βεβαίως εάν προσπαθήσουμε να νομοθετήσουμε υπερβολικά ενδεχομένως να διαραγεί αυτή η σχέση. Συμφωνώ ότι στο σύνολό της η οικονομία υφίσταται, ε, επηρεάζεται μάλλον από την ψηφιακή ενία αγορά, αλλά εμείς θέλουμε να εστιαστούμε στην οικονομία ε, γιατί θεωρούμε ότι είναι το πρώτο στοιχείο και το πιο σημαντικό και άλλωστε δεν έχουμε τη δυνατότητα εδώ να ασχοληθούμε με όλες τις πτυχές. Είναι πολύ σημαντικό να ε, καταλάβουμε ότι ε, υπάρχουν σύνορα, ε, μπορεί να μην σταματούν οι ίνες και οι γραμμές ας πούμε επικοινωνίας, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν σύνορα, υπάρχουν διαφορετικοί νόμοι, αυτό θέλουμε να αντιμετωπίσουμε δεν είναι απόλυτα σωστό ε, ε, να συγκριθούν ε, οι τηλεπικοινωνίες for example Viber and WhatsApp uh, με τις OTT over the top γιατί δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα και δεν μπορεί να υπάρχει πλήρης φορητότητα. Ωστόσο, συμφωνώ ότι δεν πρέπει να καθυστερήσουμε την ψηφοφορία γιατί όπως είπαν και πολλοί συνάδελφοι πρέπει ε, να ακολουθήσουμε το βηματισμό της Κομισιόν. Τέλος. Δεν συμφωνώ με ένα μικρό κείμενο ή ένα πολύ μεγάλο κείμενο αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν πρέπει να χάσουμε την εστίασή μας. Δηλαδή να μην βάλουμε τα πάντα στο κείμενο γιατί στο τέλος δεν θα λέμε τίποτα. Θα τελειώσω λέγοντας αυτό που είπε και ένας συνάδελφος. Δεν θέλουμε ε, φρούριο Ευρώπη ε, στην ψηφιακή ε, κοινωνία. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ κυρία μου λέει ο Πρόεδρος. Υπάρχουν βέβαια κάποιες ε, διαφορές ε, μεταξύ σας. Έρχεστε από διαφορετικές επιτροπές και βλέπετε το θέμα από διαφορετική γωνία. Θα μπορούσα να προτείνω κάτι το οποίο θα, με το οποίο θα μπορούσατε να συμφωνήσετε. Χρονοδιάγραμμα. 1η Δεκεμβρίου του 2015 και για τις δύο επιτροπές κοινή συνεδρίαση των επιτροπών για τις τροπολογίες. 14 Δεκεμβρίου ψηφοφορία στην Επιτροπή και η 21 Ιανουαρίου η ε, τελική ψηφοφορία. Βλέπετε εδώ μπορείτε να συμφωνήσετε και οι δύο. Έχουμε 100% συμφωνία. Τέλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την απίστευτη, τρομερή, υπέροχη εργασία και την επίσης τρομερή και υπέροχη συνεργασία μεταξύ σας. Κυρία Συμπρόεδρε, Ευχαριστώ. Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ε, οι συζητήσεις αυτές και οι τοποθετήσεις που ακούσαμε ε, σήμερα το απόγευμα. Συμφωνώ και εγώ ότι θα πρέπει να κινηθούμε ε, γρήγορα και να κάνουμε την ψηφοφορία πριν από τα Χριστούγεννα. Μία τεχνική παρατήρηση, γιατί έχω δουλέψει και στην Ήτρε και στην Ήμκο τώρα τίνουμε να έχουμε διαφορετικές, λίγο διαφορετικές ε, ε, πρακτικές όσον αφορά την ψηφοφορία των ε, συμβιβασμών. Ίσως να έχουμε ψηφοφορία ρήτρας 5, χωριστές ψηφοφορίες κατά τμήματα, τμήμα 1, τμήμα 2. Στην Επιτροπή Ήτρε ενδεχομένως λένε 5-1, 5-2, 5-3 ή ABC και ε, ίσως δεν θα είναι εύκολο να έχουμε χωριστές ψηφοφορίες ή έχω ψηφοφορίες κατά τμήματα στα, στις συμβαστικές τροπολογίες. Ενδεχομένω λοιπόν να, θα έπρεπε να επιλέξετε μικρότερης, μικρότερου να διασπάσετε τι συμβιβαστικές τροπολογίες ή να διασπάσετε τις, τις συμβιβαστικές σε διάφορα τμήματα έτσι ώστε η κάθε ομάδα να πει τι θέλει και να μπορεί να ψηφίσει ένα διαφορετικό τμήμα. Αυτό πρέπει να το προβλέψουμε όταν έχουμε πολλές τροπολογίες και όταν θέλουμε να περάσουμε από καθαρά διπρωματικές δημοκρατικές συγγνώμη διαδικασίες. Συμφωνείτε λοιπόν για την τροπολογία και ενδεχομένως ε, τη συμβαστική και μετά ε, να μπορούν να υπάρχουν διαφορετικά τμήματα ας πούμε σε αυτή την ε, ψηφοφορία έτσι ώστε να γίνει σαφές και σε όσους μας παρακολουθούν απ' έξω ότι προχωράμε μέσα από καθαρές δημοκρατικές διαδικασίες. Ε, βέβαια μπορούμε να ζητήσουμε και την γνώμη της γραμματείας, αλλά νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να εξηγήσουμε καλύτερα σε όλους ε, με ποιον τρόπο ε, προχωρούν τα πράγματα στο, στο κοινοβούλιο μας. 1η Δεκεμβρίου η επόμενη κοινή μας συνεδρίαση. Α, θα ανοίγουμε και το πρώτο παραθυράκι με το σοκολατάκι στο ημερολόγιο των Χριστουγέννων. Πρόεδρος Μπούζεκ, οπωσδήποτε χρειαζόμαστε ευελιξία. Τώρα μπορεί ο ένας να λέει 11A, 11B, 11C, ο άλλος να λέει χωριστή ψηφοφορία ABC, αλλά με πάση περιπτώσει στην ε, Ήτρε εμείς ε, δουλεύουμε και με τις προσθήκες. Δηλαδή μπορούμε να προσθέσουμε στο τέλος ε, δύο λεξούλες ε, ή μία ε, μικρή φράση. Δεν είναι ακριβώς συμβαστική τροπολογία, αλλά μία μικρή προσθήκη ας πούμε. Περιμένουμε λοιπόν ευελιξία που θα πρέπει να τη δείξουν και οι γραμματείες μας που θα προετοιμάσουν τους καταλόγους ψηφοφορίας. γιατί είναι η δουλειά σας συγκλονιστική όπως έχω πει επανειλημμένα και επομένως θα πρέπει αυτά τα τεχνικά στοιχεία να μας εμποδίσουν. Ευχαριστώ.